What, There's one, one place for me na Ο πρόεδρος, καθίστε παρακαλώ, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Παρακαλώ, καθίστε. Ladies and gentlemen, take a seat. Καθίστε ξαναλέει ο πρόεδρος, κυρίες και κύριοι. Αρχίζει η συνεδρίαση. Στα πολωνικά. Συνεχίζουμε την ε, συνεδρίασή μας, Στα δε πρακτικά της 11ης Τρίτου και τα σχετικά κείμενα υπάρχουν διαθέσιμα.